Αυτό θα αποκρισταλωθεί στο τελικό κείμενο και ελπίζουμε έτσι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων και κυρίως του Ευρωκοινοβουλίο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πέρα στις συζητήσεις. Λοιπόν, τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει τις προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέμα πρώτο τα βιομετρικά διαβατήρια. Δίνω το λόγο αμέσως στο συντάκτη, τον κύριο Κοέλιο, που έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Μάλστρομ, αγαπητοί και αγαπη... αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κανονισμός 2252 που υιοθετήθηκε το 2004 ήταν σημαντικός για τη βελτίωση και εναρμόνιση των προδιαγραφών των σχετικών με τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχουμε εισαγάγει ταυτοποίηση βιομετρική ε, που επιτρέπει μια αντιστοιχία ακριβέστερη των στοιχείων αλλά δεν αρκεί να μιλάμε αποκλειστικά για τα διαβατήρια Όλη η διαδικασία είναι σημαντική. Έχουμε πρώτα την παρουσίαση των εγγράφων για την έκδοση του διαβατηρίου. Εν συνεχεία υπάρχει η συλλογή των βιομετρικών στοιχείων και μετά η επαλήθευση στα σύνορα. Ε, δεν έχει νόημα να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας των διαβατηρίων αν ταυτόχρονα επιτρέπουμε να υπάρχουν άλλα αδύνατα σημεία στην αλυσίδα της όλης διαδικασίας. Παραδείγματο χάρη αυτό που ακούστηκε τελευταία, ότι 10% των βιομετρικών διαβατηρίων που κυκλοφορούν στη Γαλλία είναι πλαστά, βάσει ε, πλαστών εγγράφων και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο υπευλήθη μια αναφορά σύμφωνα την οποία 20% των δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν μπορούσαν να λεχθούν ότι είναι ακριβή η ελευθερία της κυκλοφορίας στο χώρο Σέγγεν είναι βέβαια μεγάλη επιτυχία, αλλά χρειάζεται και ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαβατήρια και έγγραφα που είναι αποτελεσματικά είναι σημαντικά. Πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα πρέπει να εδράζονται επί τη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων. Δεύτερον, χρειάζεται αξιοπιστή όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα που σχετίζονται με την ηλικία για τα παιδιά και του ηλικιωμένου ανθρώπου. Τρίτον, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα έγγραφα που χρησιμεύουν την έκδοση διαβατηρίων. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Μετά, πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται τα δακτυλικά αποτυπώματα το Συμβούλιο θα πρέπει να αποστείλει ένα ερωτηματολόγιο προς τα κράτη-μέλη που θα επιτρέψει μια ανάλυση ενδεχομένων κενών που υπάρχουν στο σύστημα ταυτοποίησης καθώς και τυχόν σφάλματα, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Αυτό έγινε κατά την αναθεώρηση του 2008 και γι' αυτό έχουμε εισαγάγει ρήτρες αναθεώρησης, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να μπορέσουμε να πετύχουμε να περιμένουμε μάλλον τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων. Ερώτηση. Έχει ήδη αποτελέσματα του ερωτηματολογίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια άλλη πρόταση, αν κάτι τέτοιο παραστεί αναγκαίο. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον άλλο συντάκτη, τον αξιότιμο κύριο Έντσου, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε τα προβλήματα που συνδέονται με τον μεγάλο αριθμό των πλαστών βιομετρικών διαβατηρίων οφείλονται πάνω απ' όλα στο ότι δεν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλο τον κύκλο που οδηγεί στην έκδοση αυτών των διαβατηρίων. Όπως είχε πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2008, το επίπεδο ασφαλείας των διαβατηρίων δεν είναι επαρκές αν ο τρόπος με τον οποίο εκδίδονται δεν είναι και αυτός ασφαλής. Εγώ πιστεύω ότι η συλλογή των στοιχείων ε, δεν είναι αρκετά αξιόπιστη. Όχι μόνο για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, αλλά εν γέννη, διότι γίνονται δεκτά έγγραφα τα οποία δεν είναι πρωτότυπα. Άρα είναι άχρηστο να εκδίδονται ασφαλή διαβατήρια αν αυτά χορηγούνται βάσει ε, ψευδών πλαστών εγγράφων θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαφή αξιολόγηση όλων των καταγραφηθισών ε, ελλείψεων στην έκδοση των διαβατηρίων και θα πρέπει να ε, τα καταγράψουμε αυτά και να επικεντρωθούμε επί της ποιότητας των εγγράφων ε, που χορηγούνται για την έκδοση διαβατηρίου. Διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά τα έγγραφα μπορούσαν να παραποιηθούν, να προστογραφηθούν πολύ εύκολα θεωρώ ότι είναι σημαντικό πρώτον να περιοριστεί ο αριθμός των εγγράφων που ζητούνται όταν χορηγείται ένα διαβατήριο. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν πρότυπα, προδιαγραφές ασφαλείας για όλα αυτά τα έγγραφα. Υπάρχει και μια άλλη εναλλακτική που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να εξετάσουμε. Θα πρέπει οι εθνικές τα εθνικά δελτία ταυτότητας να είναι τα ίδια σε όλα τα κρατη της τη Ευρωπαϊκή ή τουλάχιστον το σχήμα τους να είναι εναρμονισμένο και η μορφή του. Έτσι τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να ταξιδεύει κανείς εντός Ευρωπαϊκή Ενώσεως θα είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει βάθος μελέτη όσον αφορά αυτόν τον κύκλο που οδηγεί στην χορήγηση των βιομετρικών εντύπων, εγγράφων. Διότι θα είναι σημαντική αυτή η μελέτη και για τα μελλοντικά συστήματα. Τα smart borders, το μελλοντικό σύστημα των εφιών συνόρων. Smart borders όπως αποκαλούνται αγγλικά. Ευχαριστώ άλλη συντάκτρια, η κυρία Έρνστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στην τελευταία τροποποίηση που ζητήθηκε το 2009, μετά από τρία χρόνια γίνεται αναθεώρηση με μελέτες. Αυτό μας βρήκε σύμφωνος ως ομάδα γιατί είχαμε επιφυλάξεις για λόγους προστασίας δεδομένων και ε, για λόγους προστασίας των βιομετρικών δεδομένων η ε, πίστη στην τελειότητα του μέσου, η υπερτίμηση του και η υποτίμηση άλλων ε, κρίκων της αλυσίδας μας προβληματίζουν. Η αντιμετώπιση των βιομετρικών δεδομένων στηρίζεται σε ένα μεγάλο σφάλμα, ότι δηλαδή αυτά είναι πλέον αξιόπιστα και δεν μπορούν να ε, τροποποιηθούν. Και αυτά όμως μπορούν να αλλάξουν. Στα παιδιά είναι διαφορετικά από ό,τι στους ηλικιωμένους. Γι' αυτό ε, χρειάζονται σοβαρές και αξιόπιστες μελέτες. Ε, πάντοτε παραποιούνται τα έγγραφα Συνεχίζουν οι παραποιήσεις των εγγράφων στην Γαλλία, την Αγγλία. Δεν είναι ε, η μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει ζημία. Τα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης διαφέρουν. Το ποσοστό σφάλματος στη Γαλλία και την ε, Ολλανδία είναι πολύ υψηλά και πάντοτε θα πρέπει να ρωτάμε σε τι χρησιμεύουν τα βιογραφικά δεδομένα αφού μπορούν να ε, παραποιηθούν αν δεν ισχύουν τα δεδομένα ε, ή αν γίνει λάθος σε προηγούμενο κρίκο της αλυσίδας, τα βιομετρικά δεδομένα δεν μας βοηθούν. Ε, λίγα λεπτά χρειάστηκαν για να παρουσιαστεί μια συγκεκριμένη περίπτωση ε, παραποίησης και πολύ ε, εύκολο ε, είναι να ε, αποκρυπτογραφήσουν τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις μελέτες και τα συμπεράσματα τα οποία συνάγονται από αυτές. Σας ευχαριστώ και άλλη συντάκτρια. Η Βαρόνι Λάτφορντ έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάρλο Σκαλιό διότι ανέλαβε την πρωτοβουλία για αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση και προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ταξιδιωτικά έγγραφα να είναι ασφαλέστερα και πάνω από μια δεκαετία προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς και οι Αμερικανοί και να μην μπορούν να βρουν παραδειράκια στο σύστημα οι εγκληματίες. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά τα βιομητρικά δεδομένα και τις θεωρίες διαβατηρίων. Και πάγια υπάρχει. Υπάρχει η αμφιβολία ότι δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι αυτό το σύστημα είναι στέγανο 100%. Ε, τελικά το σύστημα είναι στεγανό πέραν της θεολογίας εάν συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι όπως πρέπει. Δεν ξέρω τα πράγματα τώρα και οι διαπραγματεύσει. ξεκίνησαν το 2009 και το Κοινοβούλιο ζήτησε και απέσπασε να μην λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα από ανηλίκους κάτω των 12. Έχουμε αυτή την συγκεκριμένη Ολλανδική μελέτη και ακριβώ είπαμε ότι δεν ωφελούν αυτά τα τεχνικά αποτυπώματα. Επίσης υπάρχει και άλλη μια μελέτη σε σχέση με τα μικροκυκλώματα και τις πληροφορίες που εκεί αποθηκεύονται. Θα πρέπει μας να μελετήσουμε, να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση και πού, ποιο σύστημα το πιο στεγανό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει μια έκθεση αξιολόγησης των ισχυουσών ρυθμίσεων και διαβατήρια και θεωρήσεις και έτσι να λάβουμε υπόψη ότι είπα έχουν ε, κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την αλυσίδα συλλογής των δεδομένων. Ας λυθεί και αυτό υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κέλλερ. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Κέλλερ που είναι άλλη μια συντάκτρια στην οποία δίνω το λόγο. Συμφωνώ με την κριτική των συναδέλφων και εγώ θέλω να ρωτήσω πού είναι η αξιολόγηση. Μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις που τέθησαν και να καθησυχάσει τις ανησυχίες μας ε, όπως τα πλαστά ε, έγγραφα στη Γαλλία και αλλού γιατί έτσι υπονομεύεται η χρησιμότητα των βιομετρικών διαβατηρίων τα οποία επίσης ε, έχουν επιπτώσεις και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Γαλλίας αναφέρει την αντισυνταγματικότητά τους γιατί υπάρχει πρόσβαση όλων στα δακτυλικά αποτυπώματα που είναι πολύ ευαίσθητα δεδομένα γιατί μπορούν να αφαιθούν κάπου χωρίς πρόθεση να αφαιθούν ε, και αυτό βέβαια ε, αμφισβητεί το ε, αν μπορούν, ε, μπορεί να εφαρμόζονται τα συστήματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι, υπάρχει το θέμα της απόπειρας πολλών αξιωματούχων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο να παίρνουμε όλα τα βιομετρικά δεδομένα των ταξιδιωτών και για ποιο σκοπό συλλέγονται τα δεδομένα αυτά. Επίσης, το κόστος τέτοιων βιομετρικών συλλογών ε, συνάδει με το όφελος που έχουμε. Υπάρχει σχέση κόστους-οφέλους θετική Πιστεύω ότι επουδενή δεν πρέπει να πάρουμε τώρα περισσότερα βιομετρικά δεδομένα και να διευρύνουμε τη χρήση τους προτού ε, δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά, σε όλες τις ανησυχίες και προτού η Κομισιόν μπορέσει να επαληθεύσει ότι ε, ε, δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλα σφάλματα στη συλλογή των δεδομένων όπως ακούσαμε για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την ευκαιρία να συζητήσει το Κοινοβούλιο το σημαντικό θέμα της ασφάλειας των συνόρων ε, με τα PNR ε, στα σύνορα. Ε, αυτό είναι σημαντικό για την ασφάλεια. Η αποτελεσματικότητα των συνόρων είναι προτεραιότητα. Το 2004 ε, ενεκρίθη ο κανονισμός για τα πρότυπα ασφαλείας με αναθεωρήσει αργότερα συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών στοιχείων στα ταξιδιωτικά έγγραφα και τις ταυτότητες. Πολλά ερωτήματα ανέκυψαν και ε, που είναι πολλά τα θέματα ασφαλείας που αφορούν το σύστημα αυτό. Ρωτώ την Κομισιόν αν η έρευνα έδειξε ότι δημιουργούνται υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας από το σύστημα, αν διευκολύνονται τα ταξίδια και αν υπάρχει καλή σχέση κόστους-οφέλους. Επίσης θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν τι πρωτοβουλίες έχει αναλάβει για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πρόβλημα της, ε, των, ε, της διασυνοριακής δόλειας ε, χρήσης αυτών των στοιχείων. Πολλά προβλήματα δημιουργούνται και από την κλοπή των διαβατηρίων. Τέλος, η τεχνολογία αλλάζει αρκετά γρήγορα ώστε τα βιομετρικά διαβατήρια να διατηρούν την εχμή τους και να ε, ανθίστανται ε, στις εξίσου ε, προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους των πλαστογράφων. Ευχαριστώ πολύ. Για τρία λεπτά η Επίτροπος Μάλμστρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η μελέτη που ζητήσατε, που εστιάζεται στα δαχτυλικά αποτυπώματα για τα παιδιά κάτω από 12 ετών διεξάγεται τώρα από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο. Το θέμα της εξοπιστίας των δαχτυλικών αποτυπωμάτων ηλικιωμένων ατόμων δεν συμπεριλήφθηκε στην εντολή, άρα δεν αποτελεί κομμάτι αυτής της μελέτης. Για να γίνει επιστημονική ανάλυση, το ερευνητικό κέντρο χρειαζόταν αξιόπιστα στοιχεία παιδιών κάτω των 12 που θα πρέπει να ληφθούν δύο φορές από το ίδιο άτομο σε ένα διάστημα δύο ετία τουλάχιστον. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να παρασχεθούν μόνο από κράτη-μέλη και η Πορτογαλία ε, δήλωσε θελόντρια να δώσει από την εθνική τη βάση δεδομένη τα διαβατήρια στοιχεία. Η πρόσβαση στα στοιχεία εγκρίθηκε από τι αρχέ Πορτογαλία τον περασμένο Νοέμβριο μετά από την ολοκλήρωση διαδικασία Πορτογαλία, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων. Γι' αυτό το λόγο η μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και τα τελικά απορίσματα δεν είναι διαθέσιμα θα υπάρξει μια διάμεση έκθεση που θα παρουσιαστεί από το Ερευνητικό Κέντρο το μήνα Μάιο φέτο. Θα παρουσιάσει προκαταρκτικά συμπεράσματα όσον αφορά την εξολόγηση των δεκλικών αποτυπωμάτων των παιδιών επί τη βάση των περιορισμένων αλγορίθμων που έχουν η πανευστημιακή αναπτύξη. Η έκθεση ενδιάμεση θα υποβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο μέχρι τον Ιούνιο που καθορίζεται από τον κανονισμό σαν προθεσμία. Τα τελικά πορίσματα θα μα δώσουν πλήρε πληροφορίε για την αξιολόγηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών κατά 12 ετών και την τεχνική εφικτότητα τη χρήση αυτών για την ταυτοποίηση και επαλήθευση. Και η τελική έκθεση επίση συμπεριλαμβάνει και μια αξιολόγηση κατά πόσο οι αλγόριθμοι για βιομετρική ταύτιση που υπάρχουν στην αγορά θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και στο μέλλον για τα δαχτυλικά αποτύπωμα των παιδιών και το σχέδιο εκθέσεω θα είναι διαθέσιμο μέσα του 2013 επί τη βάση αυτών των αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σχετικέ τροπολογίε του κανονισμού. Τώρα, όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με, την, με βιομετρική καταγραφή στοιχείων, αυτό βασίζεται σε απόφαση του περασμένου Αυγούστου που τροποποιήθηκαν οι τεχνικέ προδιαγραφέ των διαβατηρίων. Σε αυτή την απόφαση, διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσει για τα δαχτυλικά αποτυπώματα ξεκαθαρίζονται με έναν οδηγό που είναι προσωτημένο στην απόφαση όσον αφορά την καταγραφή. Θεματοφύλακα των συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει ότι συμμορφώνονται τα, διαβατήρια των κρατών μελών μόλι προδιαγραφέ. Και δοκιμάζει τη συμμόρφωση. Διεξάγεται από εθνικά εργαστήρια. Και το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο έχει ήδη κάνει συμπληρωματικέ δοκιμέ όσον αφορά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα του ηλεκτρονικού διαβατηρίου επιθελοντική βάση. Είναι ο μόνο τρόπο με τον οποίο προχωρήσουμε, διότι κάποια κάτι μέλη συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θελοντικά. Και άλλε εκθέσει επίση θα εκδοθούν τον Μάιο φέτο. Συμπληρωματικέ εκθέσει για τη συμμόρφωση του Ολλανδικού δείγματο. Εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται αναλόγω. Επίση, ετοιμάζεται μια έκθεση για την κλοπή ταυτοτήτων. Αυτό είναι κάτι που το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και όσον θα είναι έτοιμη αυτή η έκθεση θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο. Όσον από το τελευταίο ερώτημα για τα αυθεντικά έγγραφα, αυτό σχετίζεται με την κλοπή ταυτοτήτων. Γνωρίζουμε ότι γίνεται αυτό του είδου η απάτη και θα ενημερώσουμε δεόντως το Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατόν για τα αποτελέσματα της μελέτης και θα συζητήσουμε μαζί σας ενδεχόμενα μέτρα προσλήψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Και τώρα, εξ ονόματος των ομάδων, εξ του ΕλΚΑ ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Θα πρέπει να δούμε τα πιθανά ωφέλη των βιομετρικών διαβατηρίων αλλά και τις σημερινές δυσκολίες και τις δυσκολίες ε, με τα έγγραφα βάσης και την έκδοση. Έχουμε πολλά τεχνικά ε, πλεονεκτήματα που μας βοηθούν στα σύνορα, αλλά πρέπει να εφαρμόζουμε και να επαληθεύουμε τη διαδικασία σωστά και πρέπει να βρούμε ισορροπία μεταξύ της ανάγκης καταπολέμησης της τρομοκρατίας στα σύνορα και την ελεύθερη διακίνηση στο χώρο Σέγγεν και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία, αλλά περιορίζει τις προσωπικές ελευθερίες και δικαιώματα γιατί χρειάζεται να δοθούν προσωπικές πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων όταν επίκειται ταξίδι. Ε, πρέπει να υπάρχει ε, δυνατότητα ταυτοποίησης μεταξύ διαβατηρίου και του προσώπου που το έχει. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την έκδοση του διαβατηρίου θα πρέπει να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν δολίως. Όπως είπε η Επίτροπος θα υπάρξει πρώτη έκθεση προσωρινή το Ιούνιο και η οριστική το 2013. Είναι σημαντικό όσοι συμμετέχουν στη διαχείριση του συστήματος να έχουν καλή εκπαίδευση, να υπάρχει διαλειτουργικότητα του συστήματος και έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια. Δεν πρέπει να υπονομεύσουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία των εγγράφων. Ούτε τα δικαιώματα των κατόχων των διαβατηρίων είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ε, σωστές ε, διαδικασίες ε, και σε ό,τι αφορά το θέμα των δακτυλικών αποτυπωμάτων στα παιδιά. Χαίρομαι που η πορτογαλική κυβέρνηση εξετάζει να παληθεύσει τις διαδικασίες σχετικά. Ευχαριστώ. Κυρία Γκυγιόμ, θέλω να χαιρετήσω την πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή, διότι με επιτρέπει να επανέλθω σε ανησυχίε που ήδη είχα εκφράσει κατά το παρελθόν σε αξιοπιστία των βιομετρικών διαβατηρίων. Είπατε τότε ότι η εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων θα επέτρεπε τη βελτίωση τη ασφαλεία των εγγράφων των ταξιδιωτικών και αυτό είναι προ υπηρεσία, εξυπηρετεί την ασφάλεια των συμπολιτών. Μια πρόσφατη έρευνα κατέδειξε ότι 10% των διαβατηρίων των γαλλικών είναι πλαστά διότι η έκδοσή τη βασιζόταν σε πολύ εύκολα να προστοποιηθούν έγγραφα, αρκεί να, ε, ε, να αντιγράψει κανεί ένα πιστοποιητικό γεννήσεω. Τότε πώ μπορούν τα, βιομετρικά διαβατήρια και τα τσιπάκια να προστατεύσουν την ασφάλειά μα. Κυρία Γκυγιόμ, πιο σιγά λέει ο πρόεδρο γιατί οι ερμηνεί δεν παρακολουθήσουν. Πράγματι. Υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να μα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύνεση για να υπερασπιστούμε την ασφάλεια πάση θυσία και όσον αφορά και συλλογή των ε, στοιχείων και να μην μειώσουμε την ευθερία κινήσεως των πολιτών και να μην χρησιμοποιούνται εκτός κοινών συμφερόντα στοιχεία που συλλέγονται. Και κάτι άλλο. Τα σκοτεινά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από μια τέτοια εξέλιξη δηλαδή σωματικά σκάνερ, ηλεκτρονικά στοιχεία, τρόποι συλλογή ε, στοιχείων μέσω λόμπι βιομηχανικών που θέλουν να προωθήσουν κάποιες τεχνολογίες με το πρόσχημα της ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Λοιπόν, φακελώνεται ο πληθυσμό έτσι, παντού στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να υπαγρυπνούμε για να σεβαστούμε την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματά του αυτά. Γι' αυτό θα επιμείνω ότι η προσφυγή στα βιομετρικά στοιχεία ίσω θα πρέπει να είναι αναλογική προ τον επιδιωκόμενο στόχο. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνε ούτω ώστε τα βιομετρικά στοιχεία να μπαίνουν στα διαβατήρια ταξιδιωτικά ε, και στα διαβατήρια που είναι μόνο απαραίτητα. Μετά, όσον αφορά την αξιολόγηση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων σε εθνικό επίπεδο, Μα κάνατε κάποιε πολύ χρήσιμε διευκρινήσει. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπονημισία, τι διάφορε εκθέσει και η πρώτη που θα έρθει νομίζω αρκετά σύντομα. Ευχαριστούμε κυρία Αγγιγιόμ. Εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων, η κυρία Ίνφελτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πολλά ακούσαμε ήδη εδώ για την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε όλα τα στάδια. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ζήτημα, την νομιμοποίηση των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια καταρχήν, διότι στην Ολλανδία ε, ένα πρόσφατο αίτημα για πρόσβαση σε έγγραφα έδειξε ότι η ε, αιτιολόγηση που δόθηκε, ε, η δόλια χρήση και πλαστογράφηση εγγράφων υπάρχει στο ε, ε, σε επίπεδο 20 ε, με 40 υποθέσεις σε μια χώρα 17 σχεδόν εκατομμυρίων. Αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί έχουμε εισαγάγει αυτό το πολύ δαπανηρό σύστημα με τις πολλές ελλείψεις, γιατί θα πρέπει να το εφαρμόσουμε όταν τόσα λίγα προβλήματα λύνει. Νομίζω ότι και αυτές τις πληροφορίες πρέπει να μας δώσει η Κομισιόν στην αξιολόγησή της. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Στανόκα από την ομάδα των Πρασίνων για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που θα γίνει τώρα, έτσι, η τροπήση του, του κανονισμού 2252. Και επίση είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο πριν από λίγο μα ε, είπε προ το ίδιο μήκο κύματο η κυρία Μάλμστρομ. Οι πράσινοι συμφωνούν το ότι έτσι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες θα περιληφθούν στο διαβατήριο και έτσι θα υπάρχουν προσθέμενη αξία και περισσότερη ασφάλεια. Δεν θα πρέπει κανείς να βρίσκει παραθυράκια στο νόμο και έτσι να εκμεταλλεύεται ή κάποια, ή κάποια κενά στην τεχνολογία. Το Δεκέμβριο το 2004 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και βλέπουμε τώρα ότι είχε αισιοπέρασε εκείνη η διαδικασία. Και ευχαριστούμε τον κύριο Κόλλιο που είναι από την πρωτοβουλία για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Επόμενη, ομιλ... Επόμενος ομιλητής ο κύριος Ζιόμπρο από την Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Το πρωί συζητούσαμε την εμπορία ανθρώπων. Συναισθηματικά φορτισμένο θέμα βέβαια ε, ένα πρόβλημα που οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα πολλές γυναίκες και παιδιά. Η ασφάλεια στα σύνορα είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία την πλαστογράφηση και παραποίηση εγγράφων. Ε, είναι ένας τρόπος αυτός για την ε, ανάσχεση ή πάυση, ε, απαγόρευση και της εμπορίας ανθρώπων. Τα βιομετρικά διαβατήρια δίνουν πολλή ελπίδα. Η έκθεση όμως δείχνει ότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε σχέση με την ε, ε, κρυπτογράφηση και τα τσίπ. Νομίζω ότι πρέπει η τεχνολογία να βελτιωθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε. Ε, δεν βλέπω τον κύριο Ζέγκεντι. Καλώς. Το 1,5 λεπτό μπαίνει στο λογαριασμό μας. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Μπουζουτήλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ιδέα εισαγωγής βιομετρικών διαβατηρίων ρίχτηκε ώστε να γίνει δυσκολότερο να προσταγραφηθούν τα διαβατήρια. Έτσι μπορούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες μας, μπορεί να ταξιδεύουν πιο εύκολα, αλλά είδαμε ότι ακόμα και τα βιομετρικά διαβατήρια αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα. Και γι' αυτό θέσαμε την προφορική ερώτηση. Την υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλαμε λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα προβλήματα και σήμερα βλέπουμε ποιες είναι ενδεχομένε ε, λύσεις. πρέπει να πω ότι η έλεγχη στα σύνορα είναι κάτι πολύ ευαίσθητο για τους πολίτες μας. Θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, η παρουσία παρανόμων μεταναστών στην Ευρώπη, καθώς και το άνοιγμα και το κλείσιμο των συνόρων μας ε, πλήττει κάποιες ευαισθησίες. Και επανειλημμένα οι πολίτες μας μας έδειξαν ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα. Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα το Κοινοβούλιο κυρίως όσον αφορά το χώρο Σέγγεν. Και έχουμε και την τεχνογνωσία ανθρώπων όπως είναι και ο Κάλλος Κοέλιο. Και έχουμε και τη Frontex. Τα βιομετρικά διαβατήρια είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της διάστασης αυτής της ασφάλειας και γι' αυτό έχουμε κάθε συμφέρον να εξασφαλίσουμε ότι είναι αποτελεσματικά τα βιομετρικά διαβατήρια και ότι δεν μπορούν να απλωσταγραφηθούν. Ε, αντιμετωπίσουμε τις εντοπιστήστες δυσκολίες που απορρέουν από τη μελέτη, τότε μπορούμε να ωφεληθούμε. Κυρίως οι τίμιοι πολίτες που ταξιδεύουν τακτικά και που σέβονται τον νόμο θα ωφεληθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. Ε, η κυρία Childers ε, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, μετά την υιοθέτηση προδιαγραφών για χαρακτηριστικά ασφαλεία βιομετρικά στοιχεία για τα βιομετρία του 2004, το πρώτο βιομετρικό διαβατήριο, ηλεκτρονικό διαβατήριο τη Ιρλανδία εκδόθηκε το 2006. Η εισαγωγή του ηλεκτρονικού διαβατηρίου έχει σαν πρόθεση να εξασφαλίζει καλύτερη προστασία κατά το πλαστογράφηση. Η προσωπική ταυτοποίηση που εμπεριείχεται στο τσιπάκι, το βιομετρικό κάθε ηλεκτρονικού διαβατηρίου, είναι κάτι που συσχετίζει με πιο βάσιμο τρόπο τον κάτοχο του διαβατηρίου με το διαβατήριο. Ήταν σωστή, έγκαιρη η εισαγωγή. Το 2010 έκανε η Ιρλανδική αστυνομία με έρευνα και έδειξε ότι 8 διαβατήρια Ιρλανδικά είχαν παραχαραχθεί από τους Ιρλανδού, η Ιρλανδική κυβέρνηση στη δολοφονία του Αχμούτ Μαμπού, του Παλαιστινίου. Πιθανότατα τα διαβατήρια τα εν λόγω ήταν παραχαραγμένα διαβατήρια που είχαν ε, εκδοθεί πριν το 2006, διότι τα βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήριά μα είναι πολύ δύσκολο να παραχαραχθούν. Τα διαβατήρια άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω επίση είχαν εμπλακεί όμω στι υποθέσει που προανέφερα. Με προβληματίζει που ακούω για άλλε αδυναμίε και για το επίπεδο τη ασφαλεία διαβατηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε άλλα κρούσματα στο μέλλον. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θα πρέπει να πάρει στα σοβαρά τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η κυρία Αντζελίλη παρακαλώ. Ευχαριστώ Προέδρε, Επίτροπε Μάλστρομ. Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων εντός και εκτός ορίων ευρωπαϊκών από πάντα ήταν μία από τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθώς και η ενίσχυση η μεγαλύτερη και η εγγύηση του χώρου αυτού, δηλαδή να υπάρχει ασφαλής χώρος. Και γι' αυτό το 2009 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση Κοέλιο που αφορούσε το βιομετρικό διαβατήριο. Σύμφωνα με την αρχή ένα άτομο, ένα διαβατήριο και τα παιδιά θα είχαν δικαίωμα να έχουν το δικό τους διαβατήριο χωρίς να πρέπει να εμφανίζονται στο διαβατήριο των γονέων τους ε, θα ήταν ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένω θα ήταν ασφαλέστερο. Είχε τη δυνατότητα να ασφαλέστερο. Αυτή η αρχή, ένα άτομο, ένα διαβατήριο, από ό,τι φαίνεται, εκ των πραγμάτων είναι μη εφαρμόσιμο ή τουλάχιστον μη ασφαλέ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. Διότι διαπιστώθηκε ότι τα χτυλικά αποτυπώματα των παιδιών που είναι κάτω των 6 δεν έχουν τέτοια ποιότητα τόσο ώστε να επιτρέπουν μια επαλήθευση αναμφισβήτητη της ταυτότητας θεωρώντας τώρα ότι τα παιδιά είναι τα, τα, τα, αυτά που εξαφανίζονται περισσότερο είναι θύματα εμπορίας ε, ανθρώπων και σεξουαλικής ε, κατάχρησης, σεξουαλικών εγκλημάτων, θα έπρεπε να γίνουν μελέτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίζεται επαρκή προστασία των ανηλίκων, ε, κυρίω ε, όσων ταξιδεύουν μόνα του. Σα ευχαριστώ επόμενη ομιλήτρια η κυρία Ματιό για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα πρώτα θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτά τα έολα επιχειρήματα σε σχέση με αυτά τα διαβατήρια τα οποία λέγεται ότι κυκλοφορούν τα πλαστά διαβατήρια που κυκλοφορούν στη χώρα μας γιατί εμείς παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά ε, ε αυτά τα, τα, τα, έγγραφα και οπότε ε, ε Οπότε και εμεί έχουμε, έχουμε θεωρήσει έγκλημα που επισύρει ένα έτο φυλάκιση και 10.000 ευρώ πρόστιμο εάν κανεί κατέχει ένα τέτοιο βατήριο. Και έτσι ε, μπορούν οι διοικητικέ αρχέ ε, να έχουν στη διάθεσή του ό,τι χρειάζονται να καταβούν τέτοιου απάντε και σε κάθε, ε, σε, σε κάθε διοικητήριο υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Και γι' αυτό το, το, το, έχουμε ενισχύσει το, το, το, το πλαίσιο ε, της χορήγησης τέτοιων εγγράφων και που επομένως κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να περιορίσουμε τις πλαστογραφίσεις. Επίσης, και κάποια πιστοποιητικά γέννησης έχουν αθωρακιστεί έναντι της απάτης. Το Υπουργείο Εσωτερικών, όλα είναι και περισσότερο προσπαθεί, με ένα ε, γραμμικό κώδικα να κατοχυρώσει επίσης και τη βεβαίωση τόπου κατοικίας. Και ε, επίση ισχύουν πάρα πολύ αυστηροί κανόνε όσον αφορά τα δικαιωτικά που κάθε φορά απαιτούνται και την υποβολή του. Την ώρα της ε, αίτηση αλλά και την ώρα της παραλαβής της ταυτότητα και του διαβατηρίου απαιτείται η, αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος. Επίση υπάρχουν ασφυρά μέτρα αντικατάσταση των κλαπέντων και απολυστέντων. Και βέβαια συνεργάζομαι και με τι αρχέ όπω με την. Τώρα τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε και με την Ιντερπολ. Ούτω ώστε να μην έχουμε χρησιμοποιήσει αυτών των ταξιδιωτικών εγγράφων ε, για σκοπού ε, παρανόμου. Και διακόπτω το μικρόφωνο. Ευχαριστούμε κυρία. Ευχαριστούμε λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα προχωρούμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πέντε ε, ε, ονόματα. Νικολάζε Κέλλη, Σέμκε, Όμπερ Μάιερ και τέλος ο κύριος Λούαν. Κύριε Νικολάζικ, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, δημιουργούνται φόβοι όσον αφορά την αξιοπιστία των βιομετρικών διαβατηρίων στην Ευρώπη. Και δεν βρήκαμε καλή λύση ακόμα. Παρόλο που χρησιμοποιούνται σε αρκετά κράτη-μέλη πάνω από πενταετία τα βιομετρικά διαβατήρια. Η αντικατάσταση των κλασικών με βιομετρικά διαβατήρια, που συμπεριλαμβάνουν ειδικό τσιπάκι με βιομετρικά στοιχεία, που είναι μοναδικό τσιπάκι για κάθε άτομο, θα έπρεπε να μας βοηθήσει να αποφύγουμε την πλαστογραφία. Όμως γίνονται εκτιμήσεις ότι ακόμα και εκατομμύρια τέτοια βιομετρικά διαβατήρια ίσως να είναι πλαστά ή να έχουν εκδοθεί βάσει πλαστών εγγράφων δικαιολογητικών. Και αυτό δείχνει ότι τα βιομετρικά διαβατήρια δεν αρκούν για να ξακριβωθεί η αυθεντικότητα των εγγράφων. Είναι θέμα που άπτεται τη εσωτερική ασφαλεία και τάξεω τη Ευρωπαϊκή Ενώσης. Άρα υποστηρίζω αυστηρότερου κανόνε που θα ισχύουν όχι μόνο για το διαβατήριο, αλλά και για τι διαδικασίε για την έκδοση αυτών. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το πρωί εδώ στο Κοινοβούλιο ε, γκρίθηκε συμφωνία μεταξύ ημών και τη Ευρωπαϊκής, ε, της, τον είπα για το PNR και αυτό θα έπρεπε να μα βοηθήσει τελικά να γίνει ασφαλέστερο το ταξίδι για όλου. Είναι ανησυχητικό που άκουσα προηγουμένω ότι 10% των γαλλικών διαβατηρίων είναι πλαστά παρόλο που ο συνάδελφος διαφωνεί. Παρόλα αυτά, παρά το, όποιο και να είναι το ποσοστό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτοί που κατέχουν πλαστά διαβατήρια πιθανότατα ε, είναι κάποιου είδους εγκληματίες. Και αν μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των πλαστών διαβατηρίων, θα κάνουμε τον κόσμο πολύ ασφαλέστερο. Επίσης και τα παραμειμένα προϊόντα, λαθρεμπόριο, ε, εμπορία ανθρώπων θα μειωθούν. Ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε συνάδελφος από την Ιρλανδία, ότι τα πλαστά διαβατήρια ήταν αυτά που ήταν πριν από τα βιομετρικά διαβατήρια. Άρα η βιομετρική τεχνολογία έχει ένα ρόλο να παίξει για να βοηθήσουμε το ώστε η κατάσταση να γίνει για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έμκε για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε, σε ευχαριστώ. Τα βιομετρικά διαβατήρια ως στόχο έχουν το πώς η ζωή των εγκληματιών θα γίνει πιο δύσκολη. Και από ό,τι φαίνεται είναι η καλύτερη δυνατή λύση την δημητρικά διαβατήρια για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Όμω, όμω, από όσο φαίνεται, τα δικαστή. και αυτά τα διαβατήρια μπορούν να πλαστογραφηθούν και όντω οι εγκληματίε μπορούν να χειραγωγήσουν τα μικροκυκλώματα αλλά και τους ε, γραμμικούς κώδικες. Σήμερα τόσο είπε η Επίτροπος θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την διαδικασία περισσότερο η Frontex αλλά και η Interpol. Ευχαριστούμε και για την τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Όμπερμαϊρ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζαμε ότι τα ε, νέα βιογραφικά, ε, τα βιομετρικά στοιχεία θα μας οδηγούσαν σε ασφάλεια, αλλά δυστυχώς ε, αναφέρεται ότι ε, είναι πλαστά ένα εκατομμύριο βιομετρικά διαβατήρια. Ε, Στη Γερμανία υπάρχουν φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα που πολλές φορές όμως ε, ε, δεν είναι αναγνώσιμα. Επίσης τα παιδιά και στους ηλικιωμένους είναι ακόμη πιο δύσκολο να ε, εξεταστούν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι λοιπόν ένα αμερικανικό δαπανηρό μέσον που δεν δίνει τα υπεσχημένα αποτελέσματα. Τώρα θα αξιολογηθεί μετά από τρία χρόνια αν ε, έχουν νόημα σε τελευταία ανάλυση τα βιομετρικά διαβατήρια. Ευχαριστώ πολύ και τέλος ο κύριος Λούαν, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα βιομετρικά διαβατήρια έγιναν αποδεκτά με δυσκολία από τον πληθυσμό εν γέννη είμαστε αντίθετοι προς την καινοτομία αν δεν εξηγείται παρκώς. Σίγουρα το σύστημα φαίνεται πολύ ασφαλές. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν οι απάτες. Διότι αυτό επιτρέπεται από την τεχνολογία και τους μηχανισμούς χάρη των οποίων οι πειρατές της πληροφορικής κλέβουν τα στοιχεία που αποθηκεύονται στο τσιπάκι. Και πιστεύει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κλέψει κανείς τα στοιχεία στο τσιπ. όπως κλέβεται και από τις τραπεζικές κάρτες. Θα έπρεπε ίσως να εξηγήσουμε καλύτερα στον κόσμο τι είναι ένα βιομετρικό διαβατήριο. Ποια μέτρα ασφαλείας συνοδεύουν αυτό το βιομετρικό διαβατήριο, ποια χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ίσως στο μέλλον θα χρειαζόμαστε ένα σύστημα ταυτοποίησης που θα χρησιμοποιεί ραδιοφωνικές συχνότητες και θα μπορούσαμε να φροντίσουμε ούτω ώστε μόνο οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να αποκρυπτογραφούν μέσω αυτών των συχνοτήτων τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Τέλος, δίνω πάλι το λόγο στην Επίτροπο Μάλμστρεμ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το εδώ πέρα μιλούμε για κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, για την ασφάλεια των ξένων εργάτων και μιλούμε για το, το, το, πόσο αποτελεσματικά μπορεί να είναι αυτά τα ταξιδιωτικά ε, έγγραφα και τα δημοτικά. Κάπω ε, άστοχο είναι το ότι σήμερα τα, τα συζητούμε. Για τον Ιούνιο θα μπορούσα να απαντήσω όλε αυτέ τι ερωτήσει και τότε θα, θα είχατε τι εκθέσει που θέλατε και τότε θα μπορούσα να σα ανακοινώσω πολλά αποτελέσματα. Τέλο πάντων, ε, ε, εγώ περιμένω πώ και πώ να τα ξαναπούμε τα εγχωριθρησκεία στα κεντρό όσον αφορά τα προστογραφημένα. Βεβαίω και γνωρίζουμε για το πρόβλημα και δεν έχω υπάρχει βεβαίωση των σχετικών ε, στοιχείων των φημών που κυκλοφορούν είναι λίγο υπερβολικές αλλά θα συνεργαστούμε με Europol και Frontex για όλα αυτά και επομένω τελικά πρόκειται να, να τα, να τα συζητήσουμε τα περί, τα περί υπεξαίρεσης κλοπής της ταυτότητας τώρα να τα βιομετρικά ε, όταν ξεκίνησε αυτή η επόμενη δεν υπήρχε ρήτρα αξιολόγηση, οπότε κανεί δεν μα είχε ζητήσει να κάνουμε τέτοια αξιολόγηση όσον αφορά την χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των βιοτερικών Και επομένω ε, αυτό το θέτει πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίω και εμεί θα πάρουμε αυτό το αίτημα υπόψη πάρα πολύ. Σα πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ σύντομα ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε και θα σα έχω να σα για μένα αποτελέσματα για τη συζήτηση. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτού του θέματος και προχωρούμε στο επόμενο που είναι προφορικές ερωτήσεις για να απαντηθούν το Συμβούλιο για την οριοθέτηση μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρώτη ομιλήτρια για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι απορώ για την απουσία του Συμβουλίου. Πάντως ευχαριστώ που δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για την οριοθέτηση. Συγγνώμη που σας διακόπτω, μου είναι δυσάρεστο, αλλά επειδή η ερώτηση απευθύνεται στο Συμβούλιο και επειδή το Συμβούλιο δεν παρευρίσκεται για να ακούσει και να απαντήσει, θα κάνουμε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα για να βρούμε το Συμβούλιο. Πού είναι. Selbstverständlich Βεβαίως, μην ανησυχείτε για το χρόνο ομιλία σας. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε όλους παρόντες όσοι πρέπει να είναι παρόντες. Λοιπόν, προφορικές ερωτήσεις στο Συμβούλιο Οριθέτηση Μειονεκτικών Περιοχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ΚΑΠ. Η κυρία Κόστινγκερ έχει πρώτη το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο που εμφανίστηκε. Πρόκειται για πολύ σημαντικό και ευαίσθητο θέμα ε, που έχει μεγάλη, και έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε τη συζήτηση αυτή απόψε μαζί.